σας δώσω μια πληροφορία στην αρχή. Συνεδρίασε προηγουμένως στο διευρυμένο Προεδρείο όπου και διανεμήθηκαν οι εκθέσεις πρωτοβουλίας. Το ΕΛΚ θα κάνει τις εκθέσεις για τη Ρωσία και την πολιτική γειτονίας. Σοσιαλιστές και δημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες την έκθεση για την ε, ασφάλεια στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ECR ε, ε Κίνα, ενεργειακή ασφάλεια Άλντε και Αφγανιστάν Ιγκούε. Εντάξει. Ωραία. Τώρα ερχόμαστε στην κανονική ημερήσια διάταξη, πρώτο σημείο. Ε, η ημερήσια διάταξη συμφωνείται, ο πρόεδρος δεν έχει ανακοινώσει. Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Μολδαβία. Ακόμα εδώ λέει Ευρωπαϊκή ε, Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας. Ο συγητής μας είναι ο συνάδελφος και τον παρακαλώ να μας παρουσιάσει τη γνωμοδότησή του. Thank you, Chair. Good morning, colleague. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλημέρα συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Με μεγάλη μου χαρά θα σας ενημερώσω για την όλη κατάσταση της επικύρωσης της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και έχει προσαρτηθεί και σχέδιο εκθέσεως στην όλη διαδικασία επικύρωσης. Πρέπει να παραδεχτώ ότι διαπιστώσαμε μεγάλο ενδιαφέρον από πλευρά συναδέλφων. Λάβαμε περίπου 99 τροπολογίες που αφορούσαν το σχέδιο εκθέσεως. Αυτό δείχνει μεγάλη συμμετοχή επιθυμία στενής και αποτελεσματικής συνεργασίας, ούτως ώστε να παραχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ως έκθεση, το εκτιμώ αυτό τα μάλλα. Και εξετάσαμε πολύ σοβαρά όλες τις ε, τροπολογίες για να ληφθούν υπόψη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τι το τρόπο το προϊόν θα είναι το άριστον. Σήμερα το πρωί διεξήχθη μια συμβουλευτική συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών συζητήσαμε τις τροπολογίες. Πλησιάζουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή τελικές τροπολογίες που θα σας προτείνουμε να τις εξετάσετε και θα σας ζητήσουμε και την άποψή σας, τη σκέψη σας και ελπίζω ότι ήδη αυτή την εβδομάδα θα έχουμε στο χαρτί την τελική τους εκδοχή. Δεν πιστεύω ότι όλες οι τροπολογίες θα ληφθούν υπόψη. Προσπαθούμε να τις ε, ομαδοποιήσουμε και να βρούμε τον καλύτερο συμβιβασμό, ούτω ώστε να εμπλουτίσουμε το σχέδιο εκθέσεως. Συνάδελφοι, οι τροπολογίες και τα σχόλια που λάβαμε πραγματικά αφορούσαν σημαντικά θέματα και σημαντικά τμήματα της εκθέσεως. Αυτό το εκτιμούμε. Γι' αυτό πιστεύω ότι τις επόμενες εβδομάδες θα είναι μια έκθεση για την οποία θα είμαστε υπερήφανοι. Και πιστεύω ότι η κοινή μας προσπάθεια θα παράγει όχι μόνο εκθέσεις μετά την επικύρωση, αλλά μια έκθεση που θα δίνει κάποιους προσανατολισμούς για τη Μολδαβία, για τις αρχές της δημοκρατίας ούτως ώστε να συνεχίσει τη διαδρομή της η χώρα προς την ε, ένταξη και τις σχετικές δραστηριότητες, ούτως ώστε να πλησιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση η χώρα. Μεγάλη προσπάθεια και το εγχείρημα. Εκτιμώ τη συμμετοχή όλων των συναδέλφων και προσβλέπω σε περαιτέρω σχόλια και τροπολογίες που ενδεχομένως υπάρχουν και μάλιστα μετά τις σημερινές συζητήσεις. Περιμένω λοιπόν τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας. Ja, vielen Dank. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Γκάλερ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω ε, τον συνάδελφο Στρεβίτσιος για το σχέδιο γνωμοδότησής του. Έχω την εντύπωση ότι διαφαίνεται μια σχετικά μεγάλη συνένεση με εξαίρεση τα άκρα ως ήθιστε. Πάντως, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρη αυτή η έκθεση, διότι η Μολδαβία είναι μια χώρα της Ανατολικής Γειτονίας, σε μια περιοχή που επικρατεί μεγάλη αστάθεια. Από τη μια έχουμε τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, έχουμε και την εμπειρία του 2008 της Γεωργίας και την παγωμένη σύραξη στην υπερδνηστερία, στο εσωτερικό της Μολδαβίας. Και σε αυτή τη χώρα λοιπόν βρισκόμαστε ε, παραμονές σημαντικών εκλογών που θα καθορίσουν και τον προσανατολισμό της χώρας. Εξού και ε, είναι καλό και χρήσιμο ως Ευρωπαϊκή Ένωση και προκειμένου ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όχι απλώς να δίνουμε τη συμφωνία μας και την ε, σύμφωνη γνώμη μας ένα ξέρω ναι, αλλά και σε μια συνοδευτική έκθεση να εξηγούμε ποιες είναι οι δικές μας απόψεις και ιδέες για το μέλλον της χώρας αυτής. Και να κάνουμε και μια προσφορά, να τίνουμε μια χείρα προς τη ε, δημοκρατία της Μολδαβίας, πώς βλέπουμε τα πράγματα. Βεβαίως, δική τους υπόθεση είναι αν θα δεχθούν αυτή την προσφορά μας. Ε, είναι σημαντικό να πούμε τώρα ότι εδώ εμείς σας προσφέρουμε κάτι, μπορείτε να το δεχτείτε ή να το απορρίψετε. Αν το απορρίψετε, δεν θα έρθουμε να σας επιτεθούμε, ούτε θα φέρουμε τίποτα ε, ένστολους εκεί, στα χακί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το ξέρουμε ε, για το πώς δρά και πώς αντιδρά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν γίνει πρόοδοι στη χώρα στις εξελίξεις, αλλά απομένουν ακόμα πάρα πάρα πολλά. Δεν είναι κράτος δικαίου η Μολδαβία όπως θα επιθυμούσαμε παντού. Υπάρχουν ακόμα κάποιες δομές οι οποίες ε, δεν είναι βιώσιμες εξού και η πρότασή μας και η προσφορά μας για γενικότερη και ευρύτερη συνεργασία στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. Είναι καλό αυτό για να ξέρει και ο κόσμος στη Μολδαβία τι προσφέρουμε εμείς και μάλιστα αυτά είναι γνωστά πριν από τις εκλογές και να μπορεί ο λαός να ψηφίσει, να επιλέξει ποιο κόμμα θέλει, τι του υπόσχεται κάθε κόμμα. Υπάρχουν οι μεν που έχουν την ευρωπαϊκή πορεία και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό ως πολιτική και κάποιοι άλλοι που έχουν άλλη προοπτική. Σε το φορά τώρα τις συμβαστικές τροπολογίες, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες ίσονο σημασία, τις οποίες θα ψηφίσουμε. Μπορεί και να συγκριστούμε στη ψηφοφορία, αλλά γενικότερα υπάρχει συνένεση. Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο Στρεμπιβίτσιους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές. Ήταν έξοχη μέχρι τώρα συνεργασία. Καρποφόρες οι συζητήσεις οι πρωινές, μάλιστα. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντικότατο μήνυμα τη συνέχιση των καρποφόρων σχέσεων μεταξύ της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Είχα την δυνατότητα στην προηγούμενη θητεία να είμαι εισηγήτρια για την απελευθέρωση από τη θεώρηση ταξιδίων για τη Μολδαβία. Ήταν πολύ επιτυχής η προσπάθεια. Και η συμφωνία σύνδεσης είναι ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την καλή έκθεση. Έχω υποβάλει αρκετές τροπολογίες για να εμπλουτίσω το κείμενο. Η Μολδαβία έχει προχωρήσει αρκετά Αναγνωρίζουμε τη φιλοδοξία της και τις προσπάθειες που κατέβαλε. Επαναλαμβάνω ότι η Μολδαβία θα πρέπει να συνεχίσει με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και οι εκλογές το Νοέμβριο θα είναι σημαντικότατη δοκιμή για την κυβέρνηση, για το λαό και για το να κινηθεί προς σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να καταπολεμηθεί η διαφθορά στη χώρα, χρειάζεται ελευθερία στα μέσα ενημέρωση, μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα, προστασία των μειονοτήτων και των ε, διαφόρων ε, των ομοφιλοφίλων. Όσον αφορά τις συμβαστικές τροπολογίες, είναι σημαντικές. Έχω ερώτηση για τη συμβαστική τρία. δεν καλύπτει την τροπολογία 38 παρόλο που αναφέρεται ότι καλύπτεται τονίζει η διατύπωση την ανάγκη δημιουργίας δικτύου ασφαλείας για εκείνους που θα είναι άνεργοι σαν συνέπειες της ε, μετάβασης αυτής. Είναι λάθος που δεν συμπεριλαμβάνεται αυτή η διατύπωση στη συμβιβαστική 3. Τα υπόλοιπα είναι εντάξει. Να αναφέρω ότι η ευρωπαϊκή προπτική για την δημοκρατία της Μολδαβίας θα διευθετήσει και το θέμα της υπερνηστερίας και απευθύνω έκκληση προς όλα τα μέρη να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις υπό τη μορφή 5 2 με πιο ενεργό συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, ελπίζω πραγματικά το Νοέμβριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εθετήσει τη Συμφωνία Σύνδεσης και να δώσουμε και σαφές μήνυμα στα κράτη-μέλη που θα ακολουθήσουν το παράδειγμα. Just very brief. Ο κύριος Γκάλερ, ε, πάρα πολύ σύντομα επ' αυτού. Λυπάμαι πάρα πολύ. Συμφωνήσαμε για τις συμβαστικές τροπολογίες. Είχατε την ευκαιρία να είστε παρόντες. Αποουσιάζατε. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα ουσίας και διαφωνούμε. Οπότε δεν μπορώ να υποστηρίξω τα όσα προτείνετε για τη συμπερίληψη ε, στην τροπολογία 38. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά έτσι είχαμε συμφωνήσει. Uh, uh, uh, Ευχαριστούμε και εμείς θα θέλαμε να συγχαρούμε τον εισηγητή για την πολύ καλή δικιά και εμείς υποστηρίζουμε την ε, σύναψη της συμφωνίας αυτής ε, με την Ουκρανία, ε, την Μολδαφία, ώστε να μπορούν ε, να πάρουν μια κατεύθυνση ευρωπαϊκή και να εξακολουθεί να υπάρχει πίεση υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες αυτές. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Λέει ότι η έκθεση ότι μπορεί η Ρωσία να θέλει να δημιουργήσει ένα διάδρομο πρώτα στην Κρυμαία και μετά προ την υπερδνηστερία ώστε να κοπεί η πρόσβαση στην. Ε, ε, ε την πρόσβαση των των Γεγκαούζων. Ε, νομίζω ότι πριν από τις ε, εκλογές πρέπει να επιμείνει στην, στον εκδημοκρατισμό ε, η Μολδαβία, όπως επίσης και στην καταπολέμηση της απάτης και του οργανωμένου εγκλήματος. Χωρίς μικρόφωνο, Πρόεδρος. Okay. Thank Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές. Στη... Εμείς ε, είχαμε ζητήσει κάποιες τροπολογίες ε, που ζητούσαν μεγαλύτερη διαφάνεια και ε, περισσότερη δημοκρατία στη Μολδαβία. Κάποιες τροπολογίες ελήφθησαν υπόψη Δύο τροπολογίες μας απασχολούν ιδιαιτέρως. Πρώτη είναι η 37. Η τροπολογία 47 για να μπορούν οι Μολδαβοί πολίτες που ε, ζουν στο εξωτερικό να ψηφίζουν, γιατί πολλοί είναι εκτός της χώρας τους ε, και θα πιστεύουμε ότι είναι δημοκρατικό να έχουν τη δυνατότητα να ε, ψηφίσουν Επίσης, ε, το δικαίωμα ψηφοφορίας ε, ε, όσων είναι επισήμως αναγνωρισμένοι ως πολίτες της Μολδαβίας. Όσον αφορά την τροπολογία 80 ως πράσινη, πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να επικεντρωθούμε και στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Κατά τη γνώμη μας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι υψή τη σημασίας, γιατί πρέπει να είμαστε πιο αυτάρκεις από ενεργειακή απόψεως ε, και πρέπει να ε, συνάδει η Μολδαβία περισσότερο με τους σχετικούς στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης την κλιματική αλλαγή. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, εν ονόματι της ομάδας μας ευχαριστώ τον εισηγητή. Η έκθεση προετοιμάστηκε πολύ καλά, είναι πολύ ποιοτική. Έλαβε υπόψη τις διάφορες υποβληθήσεις προτάσεις όπως ακούσατε υπάρχουν πολλές τροπολογίες. Εγκρίνω και την όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε και τον τρόπο με τον οποίο καταλήξαμε στις συμβαστικές τροπολογίες. Πολύ καλή δουλειά έγινε. Υπήρχαν προτάσεις των συναδέλφων στην ομάδα μας που δεν ελήφθησαν υπόψη. Δεν ελήφθησαν υπόψη όλες. Εν ονόματι του συμβιβασμού θα υπερψηφίσουμε την έκθεση. Πιστεύουμε ότι η Μολδαβία χρειάζεται το μήνυμα που θα στείλουμε μέσω της εκθέσεως πρέπει να τους πούμε ότι η πόρτα μας είναι ανοιχτή και το επόμενο βήμα θα είναι η γεωργία. Χρειαζόμαστε παρόμοια έκθεση για τη γεωργία και παρόμοιο μήνυμα που θα αποσταλεί προς τη γεωργία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα λέμε ότι είμαστε ανοιχτοί προς αυτούς, ότι είναι πρόσδεκτοι και ότι θα θέλαμε η γεωργία να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχει προοπτική προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πύρος Πρόεδρε. Δυστυχώς δεν είχα τις συμβαστικές ε, πριν τη συνεδρίαση. Σήμερα το πρωί συζητήθηκαν, οπότε δεν μπόρεσα να εξετάσω εις βάθος τις συμβαστικές. Εν πάση περιπτώσει, έχοντας διαβάσει όλες τις τροπολογίες που κατετέθησαν, πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε τρόπο ούτως ώστε να αναφέρουμε το ότι ο Πρωθυπουργό της Δημοκρατίας της Μολδαβίας ανακοίνωσε επισήμως ότι το 2015 αυτή η χώρα θέλει να καταθέσει έτοιμα υποψήφιας χώρας. Α, δεν υπάρχει όμως αναφορά στο έξοχο κείμενο του κ. Στρεβίτσιους ούτε στις τροπολογίες αυτή η αναφορά. Δεν αναφέρεται αυτό γεγονός. Δεν μπορούμε να τα γνώμε παντελώς αυτή την πολύ επίσημη δήλωση του Μολδαβού Πρωθυπουργού Κάτι που επαναλήφθηκε και από την κυρία Γκέρμαν, την Υπουργό Εξωτερικών. Δεν μπορούμε να υποκρινόμαστε ότι δεν συμβαίνει κάτι. Θα πρέπει να το αναφέρουμε ότι σημειώνουμε το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργό της Μολδαβίας αναφέρει αυτό το πράγμα. Είναι σημαντική χειρονομία. Δεν είναι κάποιο σχόλιο, κάποιο δημοσιογράφου που ακούστηκε ή οποιοδήποτε πολιτικού ανθρώπου. Είναι ο Πρωθυπουργό της χώρας που το ανακοινώνει αυτό για τον επόμενο χρόνο. Πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να γίνει πριν άλλη έκθεση ε, του Κοινοβουλίου συνταχθεί για τη Μολδαβία. Καλό τους συναδέλφους να βρουν έναν τρόπο ούτω ώστε σε συμβαστικό κείμενο ή μέσω προφορικής τροπολογίας παραδείγματος χάρη να γίνει αναφορά αυτού του επίσημου αιτήματος της επίσημης ανακοίνωσης του Πρωθυπουργού. Ευχαριστώ. Thank you. I uh, Ευχαριστώ και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, εξαιρετική του έκθεση. Είχα ζητήσει να προσθεθούν κάποια στοιχεία που μπορούν κατά τη γνώμη μου να συνεισφέρουν στην ε, πολύ καλή βάση που μας ε, έχει δώσει ο ε, αλλά είχαμε κάνει κάποιες συζητήσει ε, στις προηγούμενες συνεδριάσεις της ε, Επιτροπής μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η έκθεση αυτή να αποστείλει ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης ενθάρρυνσης στους Μολδαβούς πολίτες και στις αρχές της δημοκρατίας της Μολδαβίας. Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος κατά την τελευταία περίοδο και νομίζω ότι είναι καθήκον μας να αναγνωρίσουμε τα επιτεύγματά τους το πολιτικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή είναι ε, αρκετά ιδιαίτερο και στη Μολδαβία αλλά και στην ευρύτερη περιοχή και το δικό μας κείμενο μπορεί να κάνει τη διαφορά όχι μόνο προς το περιεχόμενό του αλλά και σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα και προς το διάγραμμα έγκρισής του. Νομίζω ότι είναι κρίσιμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει περαιτέρω προσπάθειες ε, επικοινωνίας, γιατί η καλή δουλειά μας δεν είναι αρκετή αν δεν μπορούμε να ε, τη γνωστοποιήσουμε τη δουλειά αυτή αποτελεσματικά στους πολίτες μας. Πρέπει να μπορούν οι πολίτες να γνωρίζουν ε, τις, τα συγκεκριμένα ωφέλη που προκύπτουν από τη σύναψη μιας τέτοιου τέτοιου συμφωνίας, γιατί συχνά Υπάρχει πολλή ε, προπαγάνδα και ε, ενόψη των ε, εκλογών και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα σε σχέση με αυτά που άκουσα από την Φεντερίκα Μογκερίνη εχθές για το θέμα αυτό πρέπει να υπάρξει μια ενημερωτική εκστρατεία για να μπορούν οι πολίτες να γνωρίζουν τα ωφέλη μιας τέτοιας συμφωνίας. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με αποτελεσματική επικοινωνιακή στρατηγική. Thank you, like to share... Ευχαριστώ. Κάποιοι συνάδελφοι και από άλλες ομάδες έχουν ε, Εκφράστηκαν στι ανησυχίε του για την υπερνηστερία. Είναι πραγματικά ε, πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τη ρωσική διπλωματία για το θέμα αυτό. Ε, εγώ αναγνωρίζω ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά, πάρα πολύ δουλειά από τον εισηγητή. Η πρώτη μου εμπειρία αφορούσε την ε, αντίστοιχη συμφωνία με την Ουκρανία. Παρά τις πολιτικές διαφορές μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλή συζήτηση, νομίζω, και μάλιστα πολύ σύντομα. Εμείς ε, δεν έχουμε ζητήσει τροπολογίες, κάτι το οποίο ε, δείχνει ακριβώς ότι είμαστε σύμφωνοι με αυτήν την συμφωνία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ε, ε, το εξής, να προσθέσω κάτι μόνο για ε, τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η νομοθεσία σε σχέση με το ευρωπαϊκό μοντέλο και τη στρατηγική για τις ίσες ευκαιρίες. Νομίζω αυτό θα πρέπει να προσθεθεί στις προτάσεις μας για να αρχίσουμε ε, και μια στρατηγική για την ένταξη των Ρωμά στην κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αποδείξουμε ποια είναι η δική μας θέση. Είναι μια ομάδα που υφίσταται διακρίσει στη Μολδαβία, κλεισμούς και πολύ συχνά τους εκμεταλλεύονται διακινητές ε, για εμπόριο οργάνων, ακόμα και για τη βιομηχανία του σεξ. Ευχαριστώ. Well, uh, <coughs> uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, για τις ερωτήσεις σας. Πρέπει να λάβουμε υπόψη στις συζητήσεις μας για τη Μολδαβία και κάποιες πτυχές. Είναι μια χώρα που υπάρχει παγωμένη σύραξης και είναι εισαγόμενη κρίση. Δεν είναι εσωτερική σύγκρουση αυτή. Δεύτερον, αλλάζει η χώρα. Διαφορετική πολιτική άποψη τώρα. Προσβλέπουν προς το μέλλον, χρειάζονται τη στήριξή μας, τη συνεργασία μας. Και καμιά φορά πολιτική και οικονομική στήριξη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παράγοντας πρέπει να ληφθεί υπόψη πριν τις εκλογές. Για 20 χρόνια η Μολδαβία ε, δεν είχε κάποια σταθερή θέση, ήταν ε, στο μέσο του πουθενά. Η ηγεσία τώρα της χώρας έχει κάποια στατηγική και φαίνεται ότι ο λαός της Μολδαβίας υποστηρίζει την αλόγω στατηγική. Υπάρχουν πολιτικές και οικονομικές πιέσεις που απομένουν και καμιά φορά έχουμε και μποϊκοτάζω μεγαλύτερες χώρες ανατολικές που δεν βοηθά αυτό την Μολδαβία να ξεπεράσει τα οικονομικά της προβλήματα. Έχουμε και διμερή υποστήριξη που παρέχουν οι χώρες μας στη Μολδαβία. Γιατί αναφέρεται υποστήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης στην όλη κατάσταση της Μολδαβίας. Λοιπόν, συγκεκριμένες τώρα τροπολογίες. Συνάδελφε Φασούν, εκεί αναφέρατε ένα κοινωνικό δίκτυ ασφαλείας ότι πρέπει να υπάρχει. Αναφέρεται αυτό στην τροπολογία μας που κάνει λόγο και παραθέτω να αντιμετωπιστεί εγκαίρως και σωστά η κοινωνική συνέπεια των διαφόρων σχετικών μεταρρυθμίσεων. Η Μολδαβία σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να έχει κάποιο κοινωνικό δίχτυ ή κάποιους πόρους που θα μπορούσαν να διατεθούν για αυτό το σκοπό. Καλούμε τη χώρα όμως να ασχοληθεί με το πρόβλημα και να προετοιμάσει δεόντως την όλη κατάσταση για παν κοινωνικό ενδεχόμενο από τη στιγμή που θα γίνουν αυτές οι πλήρες μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται και αυτή η τροπολογία νομίζω ότι λαμβάνεται σωστά υπόψη στις συμβαστικές προτάσεις. Ο Τσάλ Τάνοκ ανέφερε τις δράσεις της Ρωσίας που στρέφονται κατά της Μολδαβίας και την όλη γεωπολιτική κατάσταση που περιβάλλει τη Μολδαβία. Συνάδελφοι, χρειαζόμαστε πιθανότατα άλλη μια πρόσθετη παράγραφο από αυτού για να λάβουμε υπόψη τις υποβληθείς τροπολογίες και την παρούσα κατάσταση. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε κάποια συμβιβαστική, σε κάποια τροπολογία αργότερα αυτή την εβδομάδα που ελπίζω να λαμβάνει υπόψη όλες τις ανησυχίες και όλες τις γεωπολιτικές εξελίξεις που έχουμε υπόψη μας. Έτσι, σωστά θα αντιμετωπίζουμε, μάλλον θα αναφέρουμε την όλη πολιτική και γεωπολιτική κατάσταση. Ο συνάδελφος αναφέρθηκε στο δικαίωμα ψήφου των πολιτών ε, στο εξωτερικό. Αυτή είναι εθνική απόφαση. Πολλά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα για τους πολίτες τους. Πώς μπορούμε να ζητήσουμε από τη Μολδαβία κάτι τέτοιο. Γνωρίζω ότι οι πολίτες της Μολδαβίας πολύ συχνά ταξιδεύουν στο εξωτερικό κυρίως για οικονομικούς λόγους. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Ας μην προτείνουμε πράγματα που δεν εφαρμόζουμε οι ίδιοι. Καλός δρόμος να ακολουθήσουμε. Εγώ είμαι υπέρ της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, αν είναι ασφαλής και εγγυάται την πρόσβαση των πολιτών μας στην κάλπη, αλλά η πραγματικότητα θα πρέπει να μας οδηγήσει προς τα μπρος, να προοδεύσουμε να μην κάνουμε ασκήσεις θεωρητικές επί χαρτού. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πρέπει να αναφέρεται αυτό. Ήδη έχουμε κάποια αναφορά στο κείμενο, αν όχι επαρκώς, δεν καλύπτει επαρκώς το θέμα, ίσως βρούμε μια καλύτερη διατύπωση. Ο κύριος Πρέντα, αναφερθήκατε στη δήλωση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών για τις προετοιμασίες της χώρας. Είναι Κάτι πρέπει να ληφθεί υπόψη, πολιτικές αποφάσεις. Εάν το Κοινοβούλιο της Μολδαβίας θετήσει αυτή την απόφαση, εγώ θα είμαι υπέρ να αναφερθεί μια θέση ή αν υπάρχει κάποια διακήρυξη, κυβερνητικό διάταγμα που αναφέρει προετοιμασία συγκεκριμένη ημερομηνία. Μ' αρέσουν οι ρητές δηλώσεις, οι προφορικές δηλώσεις, δείχνουν πολιτική βούληση, αλλά χρειαζόμαστε έγγραφο κάτι συγκεκριμένο, κάτι επίσημο, εγκεκριμένο για να μπορούμε να αναφέρουμε αυτή την απόφαση σωστά. Βέβαια, καταλαβαίνω και εκτιμώ τι δηλώσει του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εξωτερικών, τους γνωρίζω προσωπικά και του εμπιστεύομαι. Είναι οι σωστοί άνθρωποι, τη σωστή εποχή που μπορούν να ηγηθούν της χώρας. Λυπούμε όμω, δεν θα μπορούσα να λάβω τη δήλωση υπόψη για την ώρα μπορεί να αναφέρεται σε μια πολιτική συζήτηση. Και είναι πολύ σωστό αυτό που κάνατε, που τα αναφέρατε. Η κυρία Πόστα αναφέρθηκε στην ένταξη των Ρωμά, στη συμπερίληψη των Ρωμά. Υπάρχει μεγάλη κοινότητα Ρωμά, πράγματι, που ζει στη Μολδαβία. Αναφερθήκατε σε εθνοτικές κοινότητες. Ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε να αναφέρουμε για μία ακόμη φορά τους Ρωμά, να το υπογραμμίσουμε το θέμα για μία φορά. Είναι πολύ ευαίσθητο πράγματι και στη Μολδαβία και στην γενικότερη περιοχή. Ίσως καταλήξουμε σε τελικές τροπολογίες που θα αναφέρονται στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ συνάδελφοι για τις παρατηρήσεις σας, για τα σχόλιά σας. Είναι κοινή προσπάθεια, κοινό εγχείρημα και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε στην επιθυμητή έκθεση. Ευχαριστώ. Στις 16 Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε και στην Ολομέλεια τον Νοέμβριο, την πρώτη Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Συμφωνούμε. Το Γεωργιανό θα το δούμε το Δεκέμβριο στην Ολομέλεια. Αυτό είναι ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός μας. Για τη Γεωργία λοιπόν... Η ΙΝΤΑ ψηφίζει σήμερα για τη Μολδαβία, Επιτροπή Εξωτερικού Διεθνούς Εμπορίου. Για να μπορέσει να τηρηθεί και το δικό του χρονοδιάγραμμα. Ερχόμαστε λοιπόν στο σημείο 6 στην ημερήσια ε, διάταξη. Πήγα να πω 7, αλλά 7 είναι ημερομηνία, 7 Οκτωβρίου. Το γράψαμε στην ημερήσια διάταξη γιατί γίνεται τώρα μια νέα συζήτηση. Ε, γιατί υπάρχουν προκλήσεις ε, που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ακούμε ότι και σε πολλά κράτη-μέλη δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση. Κατά τα άλλα, τον Ιούνιο, αν δεν απατώμε, του 2015 θα διεξαχθεί μια νέα σύνοδος κορυφής που αποφασίστηκε το Δεκέμβριο του 2013 στο ε, ε, Σύνοδο Κορυφής για θέματα αμήνης. Και νομίζω ότι είναι έγκαιρη τώρα αυτή η ε, προσπάθεια να ασχοληθούμε με το θέμα. Επίσης σήμερα το πρωί αποφασίσαμε να κάνουμε έκθεση για το θέμα της ασφάλειας ευρύτερα Οπότε ε, πρέπει τώρα να μας απασχολήσει αυτό το θέμα. Δεδομένων των δυνατοτήτων που έχουν στους προϋπολογισμούς τα κράτη-μέλη, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε φτάσει σε κάποια όρια στις αμυντικές δαπάνες. Και αυτά είναι πράγματα που δυσκολεύουν πάρα πολύ και τις ένοπλες δυνάμεις και γενικότερα τα θέματα ασφαλείας. Το κόστος της μη Ευρώπης στην έρευνα και μόνο στην έρευνα σημαίνει ότι αν υπάρξουν ευρωπαϊκές δομές μπορούμε να έχουμε οικονομίες της τάξεις των 26 δισεκατομμυρίων ευρώ. 26 δις. Αυτά τα έχει υπολογίσει η Επιστημονική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή, δεν θέλουμε περισσότερα λεφτά για την άμυνα, αλλά καλύτερα να πιάνουν τόπο τα χρήματα που έχουμε με συνέργειες, με συνεργασίες, με ευρωπαϊκή προσπάθεια. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλές εκθέσεις προς την κατεύθυνση αυτή και της ΑΦΕΤ και της ΣΕΝΤΕ και χαίρομαι που είναι εδώ ο κύριος Έλερ, αναπληρωτής ε, πρόεδρος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας. Οι εκθέσεις Ντανζάν και Γκάλερ της τελευταίας αιτίας έπαιξαν ρόλο και νομίζω θα πρέπει να αρχίσει σήμερα η συζήτηση για να το ξαναφέρουμε στο επίκεντρο της συνειδητοποίησής μας και να προχωρήσουμε όπως πρέπει. Θα παρακολούσα λοιπόν πρώτα τον κύριο Ντανζάν να μας κάνει μια σύντομη εισαγωγή, μετά τον κύριο Γκάλερ και μετά τον κύριο Έλερ και θα ακολουθεί η συζήτηση. Κύριε Ντανζάν, έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η υποψήφια, είπατε, η εκπρόσωπος το ανέφερε και χθε ε, στην ακρόασή της. Η πολιτική ασφάλειας και άμυνας Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης έχει εγγραφεί στις συνθήκες, στις ομάδες της πολιτικές μας, αλλά και στα κράτη-μέλη υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις σε σχέση με τη δομή ε, των, ε, της άμυνας αυτής της ευρωπαϊκής. Είναι πολύ πλούσιες συζητήσεις αυτές, όμως υπάρχουν και συνθήκες που πρέπει να τις εφαρμόσουμε και σε αυτές τις συνθήκες υπάρχουν πολλά άρθρα τα οποία είναι αφιερωμένα στην κοινή ευρωπαϊκή ε, πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Ε, μεταξύ της διατύπωσης βέβαια που υπάρχει στις συνθήκες και της πραγματικότητας υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα που κατά την άποψή μας και όταν λέω τη δική μας άποψη εννοώ της πλειοψηφίας ε, του Κοινοβουλίου μας βάσει της έγκρισης συνθήκης στην προηγούμενη κοινοβουλευτική ε, έκθεση σχετική στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Ε, υπάρχουν ε, αντιθέσεις όσον αφορά το επιχειρησιακό κομμάτι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σοβαρές δυσκολίες ε, για αποστολές πολιτικού χαρακτήρα ή στρατιωτικού χαρακτήρα που να είναι κατάλληλες σε σχέση με τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Να σας πω ένα παράδειγμα την Ουκρανία, τη, Λιβύα, τη Λιβύη, ε, τη Συρία και το Ιράκ. Ε, Κανένα από αυτούς τους πολέμους ε, στο περιβάλλον μας δεν έχουν βρει σωστή απάντηση στο πλαίσιο της κοινή άμυνας και ασφάλειας. Κατά τη γνώμη μου οι προσπάθειες που έγιναν στη Λιβύη ή εκτός Λιβύης είναι μια παταγώδης αποτυχία. Για την Ουκρανία Έχουμε μία, ε, κάνουμε μια προσπάθεια που βασίζεται σε κάποιο είδους μεταρρύθμιση ε, της ε, της κοινή ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας, όμως δεν νομίζω ότι είναι η κατάλληλη. Είμαστε εντελώς απόντες, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε πραγματικές κρίσεις έχουμε ε, κάποια μέσα διαχείρισης κρίσης, αλλά συνήθως εκ των υστέρων, κατόπιν εορτής. Δηλαδή προσπαθούμε να βοηθήσουμε σε ανθρωπιστικό επίπεδο μετά τις συγκρούσεις, αλλά όχι για την πρόληψη ή για τη διαχείρισή τους όταν συμβαίνουν. Υπάρχει λοιπόν αυτή η διάσταση μεταξύ του δόγματός μας, ε, των μέσων μας και, την, και της πραγματικότητας. Ε, υπάρχει και θέμα ε, ικανοτήτων. Είναι κάτι το οποίο το είπατε κι εσείς, ότι σε μεγάλες χώρες μέλη ε, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και να αναγνωρίζονται προβλήματα σοβαρά ε, προϋπολογισμού ε, και καταλληλότητας του εξοπλισμού και των υλικών. Ε, σήμερα, για παράδειγμα, πλήττεται η Γερμανία σε σχέση με την διαθεσιμότητα των, του εξοπλισμού. Είναι κάτι το οποίο μόλις ήρθε στο φως τη δημοσιοτητα και είναι πραγματικά ανησυχητικό και αφορά όλες τις χώρε Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Είναι κάτι το οποίο το είχαμε πει από τις αρχές Σεπτεμβρίου. δεν θα ανατραπεί αυτή η τάση, ούτε θα υπάρξει σταθεροποίηση δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Όσον αφορά τη διατήρηση δηλαδή το, του εξοπλισμού ε, και τη διαθεσιμότητά του ε, είναι πολύ κακά τα σημάδια που βλέπουμε. Ε, κάποιες χώρες κάνουν, κάνουν μερικές προσπάθειες, αλλά η προσφυγή σχεδόν συστηματικά σε κάποιες χώρες ε, για αποστολές ε, ανθρωπιστικές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βαρύνουν περισσότερο τις πιο προχωρημένες χώρες, για να το πω έτσι, μεταξύ των οποίων και η δική μου χώρα, η Γαλλία, η οποία εκ μέρους των 28 κάνει κάποιες προσπάθειες ε, συγκεκριμένα στην Αφρική, ενώ το σύστημα του κοινού προϋπολογισμού δεν ε, δίνει τη δυνατότητα να καλυφθεί αυτό το κόστος ε, προς όφελος όλων αυτή τη στιγμή. Λοιπόν που μιλάμε ε, για κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια πρέπει να πω ότι η γεωμετρία αυτής της δομής είναι πάρα πολύ μεταβαλλόμενη και δεν βλέπω να υπάρχουν προτάσεις οι οποίες θα αλλάξουν τα πράγματα μέσω πρόθεσμα ε, ή βραχυπρόθεσμα. Γι' αυτό ακριβώς ε, ε, είπαμε να μιλήσουμε για, το, για τη συνέχεια από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2013, γιατί τότε γνώριζαν τα κράτη-μέλη πολύ καλά την εξέλιξη του στρατηγικού πλαισίου, όπως επίσης και τα θέματα προϋπολογισμού και τα προβλήματα με τις διάφορες εταιρικές σχέσεις και τις συμμαχίες μας. Είναι κάτι που το συζητήσαμε στο Συμβούλιο και το έχουμε πει πολλές φορές και εδώ. Ε, πρόκειται για, φιλόδο, για στόχους ε, αρκετά ε, μετριασμένους και όχι πάρα πολύ φιλόδοξους. Σίγουρα δεν είμαστε στο ύψος των περιστάσεων και το γεγονός ε, ότι τον Ιούνιο του 2014 έπρεπε να ξαναμιλήσουμε για αυτό ε, το θέμα, ε, συγγνώμη, τον Ιούνιο του 2015 ε, πρόκειται να ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα. Βλέπουμε όμως ότι μέχρι τότε υπάρχει όλο και λιγότερο ενδιαφέρον γιατί δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα που να αλλάζει τα πράγματα ούτε σε βιομηχανικό επίπεδο ούτε σε επιχειρησιακό επίπεδο κάτι το οποίο να, μας, να μπορεί να δείξει στους πολίτες μας ότι ε, οι Ευρωπαίοι έχουν καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα και ανησυχούν για την άμυνα της Ευρώπης. Όταν διαβάζω τα στάδια ε, της σε προόδου ε, σε σχέση με τα συμπεράσματα που ελήφθησαν στο Συμβούλιο του 2013, έχουμε πάρα πολλή δουλειά ακόμη για ένα Συμβούλιο το οποίο ήδη δεν είχε θέσει πάρα πολύ ε, φιλόδοξους στόχους. Είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε εδώ και πολύ καιρό, ε, συνεχώς κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου, καλά κάνουμε. Οι υπεύθυνοι βρίσκονται στις πρωτεύουσε και για το καλύτερο και για το χειρότερο. Εγώ είμαι ρεαλιστής και συνειδητοποιώ ότι τα κράτη-μέλη πρώτα πρέπει από επιχειρησιακή απόψεως και δημοσιονομική απόψεως να αναλάβουν τις ευθύνες που τους βαρύνουν. Ε, δεν λέω ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια ευρωπαϊκή πολιτική η οποία θα ε, προσπαθούσε να συγκεράσει πράγματα που δεν είναι δυνατόν να συγκεράσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να έχουμε κάτι το οποίο να είναι βιώσιμο ε, δεν βλέπουμε κανένα ε, πρόγραμμα που να μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, που να υπόσχεται κάτι διαφορετικό, ούτε σε επίπεδο ικανοτήτων, ούτε σε επίπεδο βιομηχανίας, ούτε σε επίπεδο επιχειρησιακό. Για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, ας πούμε, ε, τα βιομηχανικά προγράμματα ε, είτε για τα επίγεια μέσα είτε για άλλα μέσα είναι πολύ περιορισμένα ε, είναι πολύ ε, μικρή ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού εξοπλισμού. Είναι μια ανταγωνιστικότητα μάλιστα που μάλλον θα μειωθεί λόγω της περιοριστικής για τις εξαγωγές πολιτικής που κάποια κράτη-μέλη έχουν ε, προβλέψει δεν φαίνονται ευίωνα τα πράγματα, είναι μάλλον απεσιόδοξα. Ίσως να υπερβάλλω λιγάκι στην παρουσίασή μου, αλλά τη χρονική στιγμή που έγινε αυτό το Συμβούλιο, το Δεκέμβριο του 2013, που επεξεργαστήκαμε τα, τις βασικές συστάσεις, ε, ένα χρόνο σχεδόν μετά η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Και μιλάω για τις απειλές που υπάρχουν ε, στο περιβάλλον μας. Ε, μερικές φορές κατακρίνουμε τα προηγούμενα χρόνια και λέγαμε ότι ήμασταν υπερβολικοί στην ανησυχία μας τα προηγούμενα χρόνια και λέγαμε ότι ε, είναι σωστό η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να αναφέρεται στη δυνατότητα ύπαρξης πολιτικής άμυνας και στρατιωτικών ικανοτήτων. Ναι, εγώ νομίζω ότι φαίνεται πια αυτή η ανάγκη να είναι πιο επιτακτική από ποτέ, γιατί υπάρχουν πραγματικά πραγματικές ε, συγκρούσεις, πραγματικές σειράξεις οι οποίες ε, θα ε, συνεχίσουν να υφίστανται. Δεν πρόκειται η κρίση ούτε στην Ουκρανία ούτε στη Λιβύη να σταματήσει αύριο. στην, στο Ιράκ η καταπολέμηση της τροποκρατίας δεν είναι πράγματα που θα τελειώσουν ως αύριο και νομίζω ότι εμείς δεν είμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Τουλάχιστον θα έπρεπε να είμαστε λιγότερο ιδεολόγοι, να είμαστε λίγο πιο πραγματιστές στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα αυτά και πρέπει να υπάρξει προόδος όσον αφορά τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεών μας, τη ταχύ ανάπτυξη ορισμένων ε, ε, ε, ομάδων και μπορεί να, πρέπει να δούμε και το πόσο χρονοβόρα είναι όλα αυτά, γιατί μερικές φορές χρειαζόμαστε πάρα πολύ χρόνο κάποια κράτη που δεν θέλουν να συμμετέχουν, εντάξει, ε, να μην συμμετέχουν, αλλά θα έπρεπε να επιτρέπουν στα άλλα... Η ομοφωνία τους δυσκολεύει τα κράτη-μέλη, αλλά θα έπρεπε κάποια κράτη-μέλη που δεν θέλουν να συμμετέχουν να μην συμμετέχουν, αλλά να μην εμποδίζουν τα υπόλοιπα να προχωρήσουν. Ε, ας κάνουμε λοιπόν σήμερα έναν απολογισμό σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2013. Ε, παρόλα αυτά το συμπέρασμά μας ε, πρέπει να είναι πραγματικά ιδιαίτερα επικριτικό και πολύ ανησυχητικό. Ο κύριος Γκάλερ, ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, θα ήθελα να καλωσορίσω οπωσδήποτε τις συζητήσεις που κάνουμε και στην Υποεπιτροπή ΣΕΝΤΕ και καλό είναι που μεταφέρεται και εδώ η συζήτηση σε μια μεγαλύτερη ομίγυρη στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Να μην περιορίζεται μόνο στα πλαίσια της ΣΕΝΤΕ, διευρύνεται κάπως η συζήτηση. Θέλω να πω ιδιαίτερα στους νέους συναδέλφους που παρίστανται ότι τις παραμονές ε, του Δεκεμβρίου 2013 ε, για τη Συνόδου Κορυφής κάναμε τη δουλειά μας και στη ΣΕΝΤΕ και στην ΑΦΕΤ. Ε, μιλήσαμε για αυτά τα ελλείμματα που έχουν συσσωρευτεί όλα αυτά τα χρόνια και για τις δυνατότητες που έχουμε. Έχουμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα, δεν είναι η πρώτη φορά. Ανέκαθεν λέμε ότι οι δυνατότητες της συνθήκης της Λισαβόνας ε, δεν αξιοποιούνται, δεν εξαντλούνται σε καμία περίπτωση. Ανέκαθεν εγώ πίστευα ότι σε θέματα ΕΠΑΑ ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας δεν πρόκειται να προχωρήσουμε ε, εκτός αν φτάσουμε όλοι στο, στα όρια μας ε, από την οικονομική στενότητα. Ε, βλέπουμε ότι και οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν φύγει από την Ευρώπη, δεν τους ενδιαφέρει πλέον στρατηγικά ε, και ε, η κατάσταση ε, διεθνώς έχει οξυνθεί πολύ. Λοιπόν, τώρα συντρέχουν και τα τρία αυτά που είχαμε βάλει ως προϋποθέσεις. Δεν έχουμε λεφτά, οι Αμερικανοί φεύγουν και γύρω-γύρω επικρατεί πολύ μεγάλο χάος. Κάθε κρίση σημαίνει και ευκαιρία και θα πρέπει να επανέλθουμε στις αποφάσεις που είχαμε λάβει παραμονές της προηγούμενης συνόδου για την άμυνα. Τότε εγώ ήμουν λοιπόν, εισηγητής για την ε, Ευρωπαϊκή ε, Βιομηχανική Βάση για την ε, Αμυντική Βιομηχανία. Στα αγγλικά αυτό λέγεται πιο εύκολα και ο πρόεδρος λέει ακούγεται και πιο ωραίο. Ναι, όντως ακούγεται και πιο ωραίο για να έχουμε την επιχειρησιακή δυνατότητα από κοινού να εξασφαλίσουμε την πολιτική μας. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχουμε ίδια αυτόνομη βιομηχανική βάση στην Ευρώπη. Να μην εξαρτώμαστε από τρίτους σημαίνει αυτό με θερμινευόμενο. Δηλαδή, να μην πηγαίνει ο καθένας να αγοράζει εξοπλισμούς όπου του αρέσει και μετά ερχόμαστε και εκπλησόμαστε ότι δεν είναι διαλειτουργικά τα συστήματα και συμβατά μεταξύ τους. Ε, υπάρχει και μια εξωτερική διάσταση λοιπόν της ΕΠΑ που θα πρέπει να συνδυαστεί με τη βιομηχανική πολιτική της Ευρώπης και την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Έχει σημασία πιστεύω κάτι που ζητήσαμε από τότε να υπάρξει μια ευρωπαϊκή απογραφή. Τι εξοπλισμούς έχει ο καθένας. Stock taking λέγεται αυτό στα αγγλικά. Τι έχουμε. Αν ξέρουμε τι εξοπλισμό έχουμε και σε ποια κατάσταση είναι το υλικό μας, τότε ξέρουμε και τι χρειαζόμαστε. Σε ποια προοπτική όλα αυτά η ευρωπαϊκή στρατηγική θα πρέπει να ε, γραφτεί ξανά από την αρχή και ενδεχομένω να γίνει και μια λευκή βίβλος. Δεν ξέρω τι μορφή θα λάβει για την ασφάλεια και την άμυνα. Να πω και πάλι για τους νέους συναδέλφους που δεν είναι μέλη ενδεχομένω στην ε, υποεπιτροπή ΣΕΝΤΕ, ασφάλειας και άμυνας, τι χρειαζόμαστε. Εναρμόνιση. Μήπως να κλείσουμε κανένα κινητό. Ναι. Ε, εναρμόνιση των απαιτήσεων συνένωση ε, της ε, ζήτησης, συγχρονισμό των προμηθειών ε, εξοπλιστικού υλικού και τελικά κοινή εκπαίδευση. Όλα αυτά χωράνε βελτιώσεις. Εάν δεν σχεδιάζουμε από κοινού και δεν αγοράζουμε από κοινού, τότε δεν πιάνουν τόπο τα λεφτά μας. Σε όλα τα υπουργεία μας, και δεν εξαιρείται καμία χώρα ή σχεδόν καμία, εν περιπτώσει, σε όλα τα υπουργεία Έχουμε αρμοδίους για τους εξοπλισμούς και οργανισμούς για τις προμήθειες των όπλων δυνάμεων που είναι σε παλιές νοοτροπίες, σε εθνικά καλόπια και ο καθένας κοιτάει τη χώρα του και δεν έχει αυτόν τον ορίζοντα, την ευρύτητα ε, του πνεύματος να δει ε, και την Ευρώπη. Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια να έχουμε αυτές τις πατάλες. Το είπε και ο Πρόεδρος, το κόστος της μη Ευρώπης και εδώ είναι τεράστιο. Υπάρχει μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πόσα δισεκατομμύρια ετησίω ε, πετάμε. Θα πρέπει να προχωρήσουμε στην πιστοποίηση και στην τυποποίηση. Τι σημαίνει αυτό. Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δεν χρειάζεται κάθε φορά να κάνουμε νέες αιτήσει για πιστοποίησεις και επίσης χρειάζεται και ασφάλεια ανεφοδιασμού. Δηλαδή, στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μιλάω καν για εξαγωγές. Να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό που χρειαζόμαστε θα το αγοράζουμε από έναν εταίρο. Εάν υπάρχει ανασφάλεια εκεί, τότε θα πάει ο κόσμος να αγοράζει αλλού. Από εκεί που ξέρει ότι θα τον εφοδιάζουν. Ε, και όχι αγορά καλής ελπίδος να δούμε πότε θα έχει η Ευρώπη αυτό το υλικό. Στην έρευνα και ανάπτυξη τα ζητήσαμε και αυτά στην έκθεσή μας. Μια παρασκευαστική δράση για την αμυντική έρευνα έχει ξεκινήσει ήδη και η Εξωτερική Επιτροπή ΑΦΕΤ συμφώνησε και η Επιτροπή Βιομηχανίας, ακόμα και η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Η ΔΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκφραστεί και αυτή θετικά. Αυτά τα πράγματα είναι επίκαιρα, έχουν ξεκινήσει, τρέχουν αυτό τον καιρό, θα μεταξελιχθούμε και ε, είμαι βέβαιος και αισιόδοξο ότι θα προχωρήσουμε και υπό την εντύπωση που μας άφησε χτες η υποψήφια αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Μογκερίνη. Τι είπε, ότι στην ασφάλεια και άμυνα πραγματικά θέλει να ασχοληθεί περισσότερο, έχει άλλο επίπεδο φιλοδοξίας, είπε χαρακτηριστικά από την κυρία Άστον και νομίζω έχει σημασία και αυτό. Για παράδειγμα, να παρακαλήσουμε τους νέους επιτρόπους να κοιτάξουν πώς εργάζεται η Task Force για την άμυνα. Θα πρέπει να αναβαθμιστεί, να το αναλάβουν οι επίτροποι. Μέχρι τώρα είναι σε επίπεδο υπηρεσιακών παραγόντων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας από τις αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θέλω να το πω θετικά, ελπίζω στην οργανωτική αναδιάταξη τώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα τμήματα και οι υπηρεσίες που ασχολούνται με αυτά τα θέματα να μην μοιραστούν αυθαίρετα σε διάφορες γενικές διευθύνσεις. Θα πρέπει να παραμείνουν αυτά τα ζητήματα και αυτές οι μονάδες σε μια, στην ίδια γενική διεύθυνση για να μην χαθούμε οργανωτικά και κατακαιρματιστούμε στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τελειώνω θα πρέπει να μας απασχολήσει αυτό το θέμα κεντρικά. Πώς θα προετοιμάσουμε το επόμενο ε, σύνοδο κορυφής για την άμυνα, τι θα ζητήσουμε η σύνοδος του Δεκεμβρίου 2013 ίσως να ήταν ε, σχετικά νωρίς εντός εισαγωγικών γιατί η κρίση της Ουκρανίας δεν είχε οξυνθεί τόσο πολύ ούτε είχαμε καταλάβει τότε ποιες είναι οι προκλήσεις ακριβώς που αντιμετωπίζουμε. Τέσσερις μήνες αργότερα η σύνοδος αν είχε διεξαχθεί θα είχε καταλήξει και σε άλλα συμπεράσματα και αποφάσεις. Εν πάση περιπτώσει έχουμε τώρα κάποια ε, βάση ε, κάποιες αποφάσεις και θα πρέπει να δώσουμε και την πολιτική όθηση για να προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Και σίγουρα το Κοινοβούλιο ε, είναι διατεθειμένο να βοηθήσει και να συνεργαστεί προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριο Σέλερ. Νομίζω οι δύο προλαλήσαντες αναφέρθηκαν στην ε, στρατηγική σημασία και στο πολιτικό επίπεδο. Εγώ θέλω να μπω σε λίγες λεπτομέρειες, πρακτικά τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Πολλά έχουν χαρακτήρα έκκλησης προς τα κράτη-μέλη και πολλά έχουν διατυπωθεί και συμφωνηθεί αλλά όχι υλοποιηθεί στα πλαίσια της ΕΠΑΑ Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλεια και Άμυνα. Τώρα, πρακτικά τι κάνουμε. Αν δούμε την τελευταία διετία έως και τριετία, τελικά, στα πρακτικά έγιναν πολύ λίγα υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στις εξαγγελίες και στις ανάγκες και τις πρακτικές, το οποίο διευρύνεται συνεχώς. Θέλω να σας πω για δύο πρωτοβουλίες. Στο Κοινοβούλιο ένα βήμα κάναμε ε, συγκεκριμένο, η συνεργασία ΣΕΝΤΕ και ΙΤΡΕ ε, για τον ορίζοντα 2020 έχουμε ε, ε, μια αποστολή πολιτική και στρατιωτική προτείνει και διατυπώσει. Δηλαδή, σήμερα ερχόμαστε να διατυπώσουμε ότι έχουμε 200 εκατομμύρια ευρώ και μέχρι και πιλωτικά προγράμματα και πολύ συγκεκριμένα συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών, βιομηχανικά έργα, project που ε, αναπτύσσουν τις ικανότητες και δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. συστήματα διαταγής και ελέγχου, command and control. Ε, πρακτικά ε, συστήματα διοίκησης και ελέγχου δεν έχουν προχωρήσει. Ε, πρακτικά επαναλαμβάνω τα προγράμματα εργασίας, τα είπε και ο κύριος Γκάλερ. Και ουσιαστικά έγινε αυτό που φοβούμαστε. Στη Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας που ήταν ένας μεσάζων έχει φύγει αυτή η αρμοδιότητα και έχει πάει στα εσωτερικά. Τώρα θα χρειαστεί άλλο ένα εξάμεινο για να γίνει αυτή η αναδιάταξη στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρόλο που έχουμε ένα ερευνητικό προπολογισμό 1,7 δι. Τώρα μέσα εκεί θα πρέπει να κινηθούμε για την πολιτική και στρατιωτική συνεργασία και ασφάλεια. Και το θέμα μας απασχολεί στην Επιτροπή ΑΦΕΤ και στην Υποεπιτροπή ΣΕΝΤΕ, αλλά θα πρέπει να δούμε, θα παραμείνουμε στις εκκλήσεις και στις προτάσεις ή θα συνδυάσουμε όλα αυτά τα θεωρητικά με πρακτικά βήματα, με τις δυνατότητες που μας δίνει η συνθήκη, ο προπολογισμό και το ίδιο το Κοινοβούλιο. Να σας δώσω δύο παραδείγματα αυτό το θέμα των μη επαδρομένων αεροσκαφών ε, είναι επίμαχο στη συζήτηση. Αλλά η δυνατότητα, η αναγνωριστική για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ σημαντική και στρατιωτικά και πολιτικά για την ασφάλεια των συνόρων. Δεν υπάρχει καμία χώρα μέλος ε, στην Ευρώπη, στα πλαίσια της και κυκλοφορίας, στην πολιτική αεροπορία, δεν μπορεί να σηκώσει ε, μη επαδρομένα αεροσκάφη, ούτε για να φυλάσει τα σύνορα τα ίδια στα σύνορα. Στον πολιτικό τομέα, επαναλαμβάνω, δεν θα μπορούσε ε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας να βοηθήσει να δημιουργηθεί νομική βάση για να μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί αναγνωριστικά ε, μη επανδρομένα αεροσκάφη στην πολιτική αεροπορία, επαναλαμβάνω. Υπάρχουν τεράστια εμπόδια για τις δυνατότητες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι θα μπορούσα να σας αναφέρω και άλλα παραδείγματα και άλλους τομείς ε, που είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι εκκλήσεις προς τα κράτη-μέλη και παρακλήσεις. Λοιπόν, θα πρέπει να τα κοιτάξει αυτά και η ΑΦΕΤ και η ΣΕΝΤΕ, ποια είναι τα συγκεκριμένα βήματα που μπορούμε εμείς να ξεκινήσουμε. Βέβαια, η γενική κατάσταση είναι δύσκολη, το είπαν και οι προλαλήσαντες, και θα έχουμε εμείς και αυτή την ευθύνη. Αλλά πέρα από αυτά, πολύ συγκεκριμένα βήματα τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους Ντεζόν, Γκάλερ και τους άλλους. Ήταν σαφέστατοι στις παρεμβάσεις τους. Ευχαριστώ και για τις πρακτικές ε, προτάσεις τους. Θυμάμαι τη σύμβαση για το μέλλον της Ευρώπης, τη συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης, από το 2002 και τούδε επαναλαμβάνονται θέσεις, αλλά χωρίς εφαρμογή των θέσεων και των προτάσεων ε, μένουμε σε τέλμα. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν για να εφαρμόσουμε συγκεκριμένες δράσεις στην πράξη. Χρειαζόμαστε περισσότερες ε, απειλές, περισσότερες καταστροφές, ακόμα και πιο κοντά από ό,τι μέχρι τώρα. Θα πρέπει να μας ε, καθοδηγούν ε, στρατηγικής φύσεως ε, σκέψης και προβληματισμού... όσον αφορά τις παρούσες ε, απειλές. Εγώ είμαι υπέρ της ειρήνης. Αλλά βλέπω ότι γύρω μας υπάρχουν προβλήματα. Ο κόσμος καίγεται και πρέπει να εξετάσουμε τι μπορούμε να πετύχουμε με ήπια δύναμη και τι με άλλα μέσα. Ευχαριστώ. Thank you. Um, Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια νέα στρατηγική ασφαλείας χρειάζεται να εφαρμόσουμε την ισχύουσα και χρειάζεται η πολιτική βούληση και αυτό λείπει. Σε όλες σε όλου του πολιτικού Σε κάποιες χώρες για λόγους ιστορικούς υπάρχει μεγάλος δισταγμό και αντίσταση και μποϊκοτάζ όσον αφορά την κοινή άμυνα και σε κάποιες πολιτικές οικογένειες όπως και δική μου, πολλοί στην αριστερά πιστεύουν ότι όταν μιλάμε για άμυνα και ασφάλεια αυτό είναι κάτι που στέφεται κάτι σε ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όχι, αφορά την ειρήνη και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το σεβασμό του διεθνού δικαίου. Αυτή πρέπει να είναι η βάση εσδήποτε δράσεως τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα. Κοιτάξτε τι γίνεται με αυτούς που κάθονται στη μέση του Κοινοβουλίου, τους Κούρδους, που ζητούν να αναλάβουμε την ευθύνη μας να τους προστατεύσουμε και χρειάζεται να έχουμε τα κατάλληλα μέσα κάτι τέτοιο και νομικό πλαίσιο και το ηθικό πλαίσιο για να μπορούμε να δράσουμε. Δεν το έχουμε, διότι πράγματι παρά τη δουλειά, παρά τα λόγια, ε, έχουμε επενδύσει ελάχιστα στην ΚΕΠΑ. Και γι' αυτό έχουμε αυτό το ξέσπασμα των αναφλέξεων γύρω μας. Κοιτάξτε, γίνεται στη Λιβύη. Ξεκάθαρο παράδειγμα παράληψης δράσης από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να κινηθεί από κοινού συντονισμένα. Το λέγαμε από την αρχή αυτό. Πηγαίναμε συχνά, συντάσαμε εκθέσεις. Συνέτασα εκθέσεις που συνέταξα. Και τα κράτη-μέλη υπέχουν τεράστια ευθύνη, διότι προφανώς δεν ήθελαν να υπάρξει συντονισμός. Και η Λέδη Άστον δεν ήθελε να σπρώξει. Δεν ήθελαν τα κράτη-μέλη. Ήθελαν όλα είναι ο συνήθω να στέλνουν συμβούλους ε, που σε κάποια γραφεία υπουργών πουλούν εξοπλισμό και λησμονούσαν τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι η προφανής απειλή που είναι μπροστά στα μάτια μας. Τρομοκράτες, δίκτυα τρομοκρατών, μαζί με συνεργασία με κλιματικά δίκτυα που δρούν σε αυτή τη ζώνη ε, όπου δεν κινείται κανείς και είναι στο κατόφλι μας αυτή. Ο Κρίστιαν Έλλας και ο Μάικλ Γκάλερ αναφέρθηκαν στην ανάγκη να είμαστε πιο αποτελεσματικοί όσον αφορά τη δαπάνη των χρημάτων για την άμυνα σε σχέση με τα μονομένα 28 κράτη-μέλη. Δεν είναι μόνο θέμα αποτελεσματικότητα, είναι και το θέμα καταπολέμηση διαφθορά. Διότι υπάρχει μεγάλη διαφθορά όσον αφορά τι προμήθειε τη άμυνα ε, στι χώρε μα. Σήμερα στη... είχαμε κυβερνητική επιτροπή έρευνα και συζητούσαμε για την πώληση γερμανικών υποβρυχίων στη χώρα μου. Στη Γερμανία υπάρχουν κάποιοι που δικάστηκαν ήδη για διαφθορά για την παροχή, ε, για την πώληση γερμανικών υποβρυχίων στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα. Δικάστηκαν στη Γερμανία αλλά όχι στην Πορτογαλία. Διότι η διαφθορά φτάνει μέχρι τα άνω κλιμάκια, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εθελοτυφλεί και δεχόταν ψέματα, παραπλανητικά επιχειρήματα της πορτογαλικής κυβερνήσεως για να καλυφθούν οι ευθύνες στη χώρα. Είναι κρίσιμο σημασία στο θέμα για όλους τους πολίτες να υπάρχει κοινή προσπάθεια για την ασφάλεια και την άμυνα στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε λοιπόν και βιομηχανική βάση που θα είναι αυτόνομη. Να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης για την καταστροφή των δυνατοτήτων που έχουμε. Για μας που έχουμε δυνατότητες στατιωτικές και δυνατότητες ασφάλειας και δυναμικό. Είναι σαφές στη χώρα μου αυτό. Στατηγική τομής. Όχι μόνο στην Πορτογαλία αλλά και άλλοι τομείς είναι στα χέρια και των Κινέζων. Και οι στρατηγικές εταιρείες στον χώρο της άμυνας και της ε, τεχνολογία τεχνολογίας είναι στα χέρια αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή πρέπει να συνεργαστούμε, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα. Αντί να το κάνουμε αυτό, κινηθήκαμε αντίθετα με αντίθετα αποτελέσματα και πρέπει να ζητήσουμε τις ευθύνες από τους ηγέτες που εφάρμοσαν πολύ εσφαλμένες πολιτικές με τα αποτελέσματα. Να πω τελικά από τη θεσινή ακρόαση της κυρίας ε, ε, Υπουργού της Αρμόδιας της κυρίας Μογκερίνη είδαμε ε, ποια είναι η θέση και ότι πρέπει να κάνουμε σωστή, να ακολουθήσουμε πολύ σωστή προσέγγιση και χρειάζεται να πιέσουμε πάρα πολύ τις κυβερνήσεις μας και χρειάζεται να αναλάβουν οι ηγέτες των κρατών τις ευθύνες τους για αυτά που έκαναν και για τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκαν όσον αφορά τα θέματα της ε, ΚΕΠΑ. Ευχαριστώ. Αλληλεγγύη και κοινή χρήση των αμυντικών μας δυνατοτήτων είναι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη αλλά φαίνεται να μην κινούμεθα με σωστή σειρά. Μιλάμε για περισσότερες αρμοδιότητες, περισσότερους πόρους, χωρίς να αναφερόμαστε στο τι ε, πρέπει να είμαστε ε, ικανοί, πού πρέπει να αποκτήσουμε δυνατότητες, γιατί χρειαζόμαστε τους πόρους. Χρειαζόμαστε κοινή υποστήριξη για να είμαστε όλοι ασφαλείς. Τον Ιούλιο φέτος, τον Ιούλιο, δήλωσε στο ψήφισμά του για την Ουκρανία ότι κάποια κράτη-μέλη για να το πω κομψά, δεν εφαρμόζουν την απαιτούμενη αλληλεγγύη. Σε στιγμές κρίσης, που δεν είναι θεωρητική και αφηρημένη κρίση, όταν έχουμε πραγματικές απειλές για την ασφάλεια των βαλτικών χωρών, της Πολωνίας και άλλων χωρών, χρειάζεται σωστή προσέγγιση. Ακούσαμε την κυρία Μογκερίνη χθε, που είναι η υποψήφια για τη θέση της ΥΠΑ του εκπροσώπου για τα θέματα αμήνης, σαν υπουργό Εξωτερικών, είπε ότι εκπροσωπεί την παρούσα, μάλλον εκπροσωπεί και την παρούσα προεδρία και θα έπρεπε να υπάρχει πολιτική υποστήριξη μεταξύ μας εάν όλα τα άλλα είναι ε, αδύνατο εφαρμοστούν. Η κυρία Μογκερίνη αναφέρθηκε σε τεχνικής φύσεως συζητήσεις για τον νότιο αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου, για κατασκευή αυτού του αγωγού, ε, ολοκλήρωση του αγωγού, αν ηρεμήσει η κατάσταση στην Ουκρανία. Δηλαδή θα κρατήσουν τελικά οι Ρώσοι στην Κρυμαία, αυτό σημαίνει. Μπορούμε να συνεργαστούμε, ε, πρέπει να δούμε τι είναι εφικτό όμως από τεχνική πλευρά και πολιτική πλευρά. Στην ε, σύγκρουση στην Γεωργία δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν την αρχή της σύγκρουσης να στείλουμε ειρηνευτικές δυνάμεις που θα ε, εμποδιζαν μια διάδοση της σύγκρουσης ίσως δυνάμεις κάποιων ουδέτερων κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να οργανώσουν ειρηνευτική αποστολή στην Ουκρανία. Δεν διαρωτώμεθα αν αυτό θα ήταν αποδεκτό ή όχι, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει να καθόμαστε να παρακολουθούμε τις διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα υπό, το, υπό τη σκιά του Προέδρου Λουκασέκο που προτείνει να στείλει ειρηνευτική δύναμη στην Ανατολική Ουκρανία θα καθόμαστε και να παρακολουθούμε. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί αντί να παρακολουθούμε τους άλλους ούτως ώστε να ενισχύσουμε την κοινή μας άμυνα. Έχω σεβασμό για τη Γαλλία που στέλνει δυνάμεις στην Αφρική. Και συμμετέχουν και κάποιοι δικοί μας στρατιώτες σε αυτή την προσπάθεια. Είναι μικρή υποστήριξη που παρέχουμε, αλλά υπάρχει μια υποστήριξη. Η κατασκευή του αγωγού South Stream ίσως θα ήταν κάτι πολύ χρήσιμο Αλλά να μην, πουλάμε, ε, πουλάμε όπλα στη Ρωσική Ομοσπονδία όταν τα πουλάμε στην ε, Ουκρανία. Χρειάζεται καλύτερη προσέγγιση όσον αφορά την κοινή αμυνά. Πρέπει να κινηθούμε συντονισμένα και να υποστηρίξουμε και τις χώρες εκείνες της Αφρικής που αντιμετωπίζουν προβλήματα και χρειάζονται τη βοήθειά μας και είναι νέες χώρες συγκριτικά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ συμφωνώ απολύτως με τα όσα είπαν οι συνάδελφοι, λέει κυρία Ντεσανές, και υποστηρίζω πάρα πολύ τα εισαγωγικά σχόλια του Αρνό Ντανζάν. Έχει απολύτως δίκιο. Αν κοιτάξουμε γρήγορα, δεν είναι τόσο δύσκολο τον κόσμο σε τι κατάσταση είναι. Κοιτάξτε πολύ γρήγορα στην πόρτα μας τι συμβαίνει στα σύνορά μας, στην Ουκρανία. Κοιτάξτε τι συμβαίνει σε δύο ώρες ή τρεις ώρες ε, απόσταση με αεροπλάνο, στη Λιβύη, στο Σαχέλ στη Μέση Ανατολή, ε, στην Εγγύης Ανατολή. Ε, ποιος δεν βλέπει την ε, φλέγουσα κατάσταση και πόσο επίγον είναι να έχουμε μια κοινή αμυντική πολιτική. Αν έρθουμε εδώ να προσθέσουμε στο διεθνές πλαίσιο και την αποχώρηση των Αμερικανών από την Ευρώπη ιδιαίτερα, γιατί έχουν στραφεί περισσότερο προς την Ασία, καταλαβαίνουν όλοι ε, ποια είναι τα προβλήματα. Έχουμε και στενότητα οικονομική στους κρατικούς προϋπολογισμούς, οπότε το ζωτικό μας συμφέρον θα πρέπει να είναι συνενώσουμε τις δυνάμεις μας και τη βιομηχανία μας την αμυντική. Αυτό συγκεκριμένα τι σημαίνει για μένα. Περνάει μέσα από τα εξή δύο. Πρώτον, θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να δράσουμε ως ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ κάποιων κρατών που το επιθυμούν της Ένωσης, αλλά αυτή η δυνατότητα δράσης θα πρέπει να χρηματοδοτείται από το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών. Γιατί όταν υπάρχει μια δράση στα σύνορά μας, είτε σε εξωτερικά θέατρα επιχειρήσεων, οι δράσεις αυτές θα πρέπει να είναι κοινέ και ε, είναι και προς το κοινό συμφέρον και την κοινή ασφάλεια των Ευρωπαίων. Οπότε δεν μπορεί κανείς να κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια και να είναι μία ή δύο χώρες που κάνουν τη δουλειά όταν πρέπει και επομίζονται και το κόστος χωρίς καμία αλληλεγγύη στη χρηματοδότηση. Και ένα τελευταίο, δεύτερον, αν θέλουμε βεβαίως να έχουμε αύριο μια κοινή άμυνα, γνήσια, είναι πήγον αλλά και χρόνια το λέμε ότι είναι πήγον. Αλλά εδώ είμαστε στο παραπέντε, πότε θα γίνει αυτή. Μια κοινή άμυνα σημαίνει κοινή εξωτερική πολιτική, κοινή όμως. Να μπορούμε για κάποια θέματα να είμαστε ενωμένοι και από κοινού να δρούμε. Σας ευχαριστώ. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούσαμε εναρμόνιση των απαιτήσεων, συγχρονισμό, ε, εντολή για τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, προηγουμένως μίλησε κάποιος συνάδελφος για το 2013 και το Συμβούλιο μεσολάβησαν το 14 ευρωεκλογέ όμως. Και το μήνυμα ποιο είναι. Ο κόσμος όλο και περισσότερο γυρνάει την πλάτη του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συμφωνία για αυτή. παντού ε, σε όλο το πολιτικό φάσμα ανησυχεί ο κόσμος για την κατεύθυνση που έχει πάρει το ευρωπαϊκό χείρημα. Έχουμε, ε, είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα ασφαλείας σήμερα το πρωί με κάποιους διαδηλωτές. Ε, είναι κάποιοι Κούρδοι εκεί και ποια είναι η προστασία τους, έχουν βάλει κάποιες κορδέλες ή ένα, ε, ένα σύστημα προστασίας ε, των κρατών μελών στο ε, ΝΑΤΟ υπάρχει το άρθρο 5 η άνταχτη απειλή μια χώρα και νομίζω ότι τα θέματα ασφαλείας και άμυνας είναι ζητήματα των εθνών, των εθνικών κρατών σε συνεργασία με τον ΟΗΕ και θα πρέπει να ακούτε περισσότερο τα μηνύματα των τελευταίων ευρωεκλογών για το που το πάει η Ευρώπη. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. απόλυτα με τον κύριο Νταζάν στην ανάλυση που έχει κάνει όσον αφορά την ε, τα τεράστια ελλείμματα στην στρατηγική και τα τεράστια λάθη που έχουν γίνει στην πρόβλεψη και στην διαχείριση των κρίσεων ε, που αντιμετώπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια και στο Ιράκ και στο ε, Συρία και στην Λιβύη και στην Ουκρανία και με τον Ίσης αυτή τη στιγμή και να τονίσω ότι ουσιαστικά ε, πρέπει να υπάρξει μια πολιτική βούληση για να εφαρμοστεί μια στρατηγική κοντά σε όλη την άλλη ανάλυση. Δεν μπορώ να το δω από μηχανική άποψη αλλά μόνο από την ε, πολιτική. Θα συμφωνήσω επίσης ότι πρέπει να βλέπουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν για πολιτική παρέμβαση και για την τεχνολογική δυνατότητα την οποία θα πρέπει να μοιράζονται όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορεί να είναι αποτελεσματική και η άμυνα, αλλά παράλληλα να βλέπουμε και τις οικονομικές δυνατότητες. Και σε αυτό το σημείο υπάρχει μια διάσταση που δεν έχει αναλυθεί και είναι αυτή των φτωχών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία πολλές φορές έχουν κατηγορηθεί ότι μπορεί να έφτασαν και στην οικονομική δυσπραγία λόγω αυξημένων ε, αμυντικών προϋπολογισμών. Και αναφέρομαι και στην περίπτωση της Ελλάδας και στην περίπτωση της ε, Κύπρου. Νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να μπαίνουν και να ζυγίζονται όταν γίνεται αυτή η αναλύση. Ο κύριος Πέτερ λέγανε μια πολύ σωστή παρατήρηση για τις νέες απειλές και για την ανάγκη να υπάρχει αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σωστά πρέπει να στηριχθεί και η Πολωνία και οι Βαλτικές Δημοκρατίες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή. Ωστόσο, επισημαίνω την ύπαρξη μιας τρομακτικής απειλής μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή είναι η Τουρκία η οποία αυτή τη στιγμή έχει σε κλειό ναυτικό αποκλεισμό την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά κανείς δεν έχει μιλήσει για αυτό το ζήτημα. Έχει εκδώσει ναύτεξ που απαγορεύουν την αυσιπλοεία και παραβιάζουν τον διεθνή νόμο με όλες τις ε, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα. Η Κύπρος που κακώς εκατηγορήθηκε σε αυτή την Επιτροπή ότι δεν είχε εναρμονιστεί με την ε, υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το ζήτημα των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας ε, αυτή τη στιγμή υφίσταται ένα τρομακτικό κόστος από αυτή την ιστορία ε, είναι στην ακτίνα δράσης του Ίσης ο οποίος την έχει και στην στόχευσή του και επιπλέον έχει να αντιμετωπίσει και τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Τουρκία. Νομίζω κύριε Πρόεδρε, νομίζω αγαπητοί συνάδελφοι ότι αν όντως πρέπει να ισχύει αλληλεγγύη σε αυτή την ε, χώρα θα πρέπει πάρα αυτά να διακόψουμε τις ενταξιακές συνομιλίες της Τουρκίας και να τις επιβάλλουμε οικονομικές και πολιτικές κυρώσεις. Διαφορετικά όλα όσα λέμε θα είναι σε ένα θεωρητικό επίπεδο μέχρι που θα έρθει η στιγμή που θα αντιμετωπίσουμε την πραγματική απειλή. Αν θέλουμε να δείξουμε ότι έχουμε στρατηγική αυτό πρέπει να είναι μια προτεραιότητα. Σας ευχαριστώ. Mr. Ευχαριστώ πολύ. Ως ε, αναπληρωματικό μέλος της Υποεπιτροπής ΣΕΝΤ είναι πολύ σημαντικό για μένα να συμμετέχω στη σημερινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ε, οι συζητήσει για την Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια έχουν ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό. Ξέρετε ότι η πολιτική αυτή απορρίφθηκε το 1954 αν θυμάμαι καλά. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε την ίδια κατάσταση που η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την εξή κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει ένα πολιτικό γίγαντα, αλλά δυστυχώ είναι νάνο από αμυντική απόψεω και από απόψεω ασφάλεια. Μιλάμε εδώ για την βούληση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεισφέρουν στην τις αποστολές και επιχειρήσεις της ε, ε, κοινή ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας. Και θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί έχουμε την εξή ε, κατάσταση. Υπάρχουν τέτοιου είδου αμυντικέ ικανότητε, αλλά δεν έχουν ενσωματωθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και μιλάω για το Eurocorps ε, ή για τι ομάδε μάχη. Ε, δεν είναι πάρα πολύ σαφέ πώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ω τώρα. Δαπανώνται τεράστια ποσά ε, για ε, όλα αυτά, αλλά δεν υπάρχει σαφή στρατηγική για το πώς θα χρησιμοποιηθούν σε πραγματικές επιχειρήσεις ε, και σε πραγματικές αποστολές, γιατί Κυρίες και κύριοι, όλες οι αποστολές και επιχειρήσεις που έχουν αναλυφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζονται και εξακολουθούν να χρειάζονται υποστήριξη του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει μία ακόμη φορά να τονίσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να μην έχει επαρκή στρατιωτικέ ικανότητες για να μπορέσει να αναλάβει ε, όπως πρέπει τις αποστολές και τις επιχειρήσεις της στο πλαίσιο της άμυνας και της ασφάλειας. Όλοι γνωρίζουμε ότι μεταξύ ασφάλειας και άμυνας από τη μία και από την άλλη της ελευθερίας, της δημοκρατίας, ε, του κράτους δικαίου, της ε, ευημερία ε, και της ε, οικονομικής ε, ασφάλειας ε, υπάρχει τεράστιο χάσμα. Δεν μπορούμε να αναπτύσσουμε το ένα χωρίς να αναπτύσσουμε το άλλο. Και βέβαια υπάρχουν πολλά που θα μπορούσε κανείς να πει μία ακόμη φορά να πω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση και να κάνω και μία πρόταση. Ίσως στις αρχές του 2015 να πρέπει να εκφωνήσουμε μία μελέτη ε, για την ανατολική την ανατολική πλευρά της, ε, ε, την ανατολική διάσταση της ε, ε πολιτικής ασφάλειας και άμυνας γιατί την Ανατολική Πτέρυγα, γιατί εκεί υπάρχουν τεράστιες προκλήσεις, υπάρχουν και νέες απειλές ε, που αφορούν ακριβώς αυτήν την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Ευχαριστώ. thank you, Ο κύριος Τάνοκ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν ήθελα να μιλήσω, γιατί ε, μέσα στην ομάδα μου είναι πολλές οι απόψεις για το κατά πόσο είναι επιθυμητή η αποτελεσματική της ΕΠΑΑ και κατά πόσο θα πρέπει να ισχυθεί ο ρόλος της ή να την αφήσουμε στην ησυχία της. Και έχουμε ακόμα ανησυχίες σε ό,τι αφορά ε, το πώς ε, θα εφαπτώμαστε με το ΝΑΤΟ, ειδικά να μην υπάρχει ε, διπλή δουλειά και επικάλυψη και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ στην έκθεσή μου αναγνώρισα πάρα πολύ το θετικό ρόλο στον Ινδικό ωκεανό ε, ε, κατά της πειρατείας στη Σομαλία ήταν κοινή δράση με τον ΝΑΤΟ και κάποια από τα χρήματα των πειρατών ε, πηγαίνανε και σε λάθος χέρια τελικά ανοίξαμε αυτούς τους διαδρόμους και ήταν πολύ καλό αυτό αλλά θέλω επ' ευκαιρία να συγχαρώ δύο κράτη-μέλη που γνώρισαν οικονομική κρίση τη Λετωνία και την Λιθουανία που τώρα ανακάμπτουν και έχουν ε, δεσμευτεί να φτάσουν στο 2% στόχο. Το ξέρω ότι μπορούμε να έχουμε pooling και sharing και φύ άμυνα και όλα αυτά τα πολύ ωραία ως έννοιες, αλλά τελικά θα πρέπει ε, στον εθνικό προϋπολογισμό να ε, βάζουμε πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Λετωνία και η Λιθουανία άνοιξαν το δρόμο, η δική μου χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο που ήδη εκεί κινείται στο 2% και η Γαλλία ε, είναι καλά παραδείγματα. Και δεν είναι υπέρ του Λουξεμβούργου που είναι και πλούσια χώρα και ε, ε, μικρή και έχει τόσο χαμηλές δαπάνες για την άμυνα. Θα πρέπει να ε, υπερασπιστούμε τον τρόπο ζωή μας και τα σύνορά μας γιατί υπάρχουν πολλές απειλές έξωθεν που θέλουν αυτά να τα επιβουλεύονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκτιμώ τη διεξαγωγή αυτής της συζήτησης ε, στην αρχή της θητείας μας και πιστεύω ότι πέντε χρόνια ίσως αρκούν για να προχωρήσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά στον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Όπω το σκέφτομαι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγαλύτερο δυναμικό και εξουσία και δύναμη από αυτή που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαν νέο αθλητή στο γυμναστήριο είναι, που τα πάει καλά στο γυμναστήριο, αλλά δεν έχει μπει στον αγώνα, σε πραγματικού αγώνε. Τα ρεκόρ του μπορεί να είναι έξοχα οι επιδόσεις του στο κλειστό γυμναστήριο, αλλά δεν ξέρει πώς θα τα καταφέρει στην πραγματικότητα, όταν θα ανταγωνιστεί με άλλους αθλητές και υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός. Συνάδελφοι, όταν ρωτάτε, ρωτάτε τους στρατηγούς του ΝΑΤΟ που ήταν επικεφαλής των αποστολών Ισάφ στο Αφγανιστάν, στην αρχή όλα τα κράτη-μέλη, οι συμμετέχοντες από τα κράτη-μέλη, είχαν πολλούς όρους που έπρεπε να ακολουθήσουν και δεν μπορούσαν να χειριστούν διάφορες επιχειρήσεις επιτόπιες σωστά. Μετά τελικά μειώθηκαν κάποιοι όρια από δωδεκάδες που ήταν σε πολύ λίγους όρους Πρέπει να προχωρήσουμε, να κάνουμε πρακτικά βήματα για να ξεφύγουμε από τις θεωρητικές συζητήσεις και να κινηθούμε επιτόπου, να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Η ασφάλεια και άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί τις αναγκαίες δομές. Ακόμα και αν έχουμε τις δομές, αυτό θα είναι κίνηση πρόληψης. Έχοντας αυτό υπόψη, ε, παρόλα αυτά κάποια κράτη-μέλη συμβάλλουν όλο και περισσότερο, ξεκινώντας με την ομάδα των προθύμων κρατών και τελικά ίσως όλοι θα συμμετάχουν στην προσπάθεια. Εάν κινηθούμε όλοι μαζί θα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε το σωστό σκοπό. Συνάδελφοι, γιατί έχει αυτή την δύναμη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι έχουμε πολλές χώρες εταίρους που είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν. Εάν δείτε τις χώρες εταίρους που συμμετέχουν σε κάποιες επιχειρήσεις που ξεκίνησαν με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δείτε ότι η τάση είναι πάρα πολύ καλή. Κανείς δεν θέλει να συμμετάσχει σε κάποιους αναποφάσεις τους. Αλλά πολλοί θα προσχωρούσαν αν ήταν αποφασιστική η κίνηση που ακολουθούσε η Ένωση. Η διατλαντική σχέση θα πρέπει να είναι ένας διευκολυντικός μοχλός και όχι περιοριστικός. Θα πρέπει αυτή τη σχέση μας με τους άλλους από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού να τη δούμε θετικά σαν παράγοντα για να αυξήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε, το δυναμικό μας και τελικά θα αυξηθεί και η προθυμία να κινούμαστε όταν αυτό απαιτείται. Ευχαριστώ. Ε, ε, Κύριε Πρόεδρε, όταν ε, έκανα αίτηση για να πάρω το πιστόλι μου, μου είπαν πει ότι άμα πάρω ένα πιστόλι μπορεί τελικά να το χρησιμοποιήσω. Ε, γιατί κάποιος που ξέρει ότι εγώ έχω ένα πιστόλι θα με πυροβολήσει. Είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει ένα στρατό που θα είναι έτοιμο σε κάποια στιγμή ε, να τον χρησιμοποιήσει ή καλύτερα ή αν δεν είναι έτοιμο να τον χρησιμοποιήσει να μην έχει καθόλου στρατό. <laughs> Τι κάνετε όταν έρθουν οι Ρώσοι όμως. Άμα καταφάσουν οι Ρώσοι τι θα κάνετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα τρία σημεία να υπενθυμίσω. Πρώτο σημείο σε σχέση με μια παρέμβαση που έγινε για το εκλογικό αποτέλεσμα του Μαΐου το ερώτημα είναι ε, αν σε επίπεδο ασφάλειας και άμυνας ε, αυτές ε, οι εκλογές που έδειξαν ψήφο δυσπιστίας ας πούμε προς την Ευρώπη σημαίνει υποχρεωτικά ότι απορρίπτουμε την κοινή ασφάλεια και άμυνα. Υπάρχουν πολλοί ευρωφοβικοί αλλά και ευρωσκεπτικιστές και στη δική μου τη χώρα. Αν υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν είναι αντικείμενο της κριτικής αυτής για την Ευρώπη, είναι η άμυνα. Ένα θέμα το οποίο ε, δεν είναι στο πλαίσιο της λιγότερης Ευρώπης και αυτό είναι η άμυνα. Οι άνθρωποι λοιπόν που κριτικάρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και λένε ότι ε, είναι υπερβολικά παρεμβατικοί ε, σε μερικά θέματα, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που μας λένε ότι πρέπει σε περισσότερο στρατηγικά ζητήματα να επικεντρωθείτε, μεταξύ των οποίων είναι η άμυνα και η ασφάλεια. Μπορώ αυτό το παράδοξο να το τραβήξω ακόμη πιο μακριά, αν θέλω, Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ε, προσεκτικοί και να γνωρίζουμε, το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, ότι μεταξύ των λιγότερο επίμαχων ζητημάτων που θα έπρεπε να ε, εξετάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η άμυνα. Και αυτό είναι ανεξάρτητο του για ποιο χώρα μιλάμε. Και στο πλαίσιο αυτό του πολλαπλασιασμού των κρίσεων είναι κάτι που οι συμπολίτε μα, ανεξαρτήτω τη απόψεώ του προ την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμερίζονται όλο και περισσότερο. Δεύτερο σημείο αφορά την βιομηχανία. Γιατί η αμυντική βιομηχανία πρέπει εμείς ως Ευρωπαίοι να είμαστε περήφανοι ε, και να γνωρίζουμε ότι έχουμε μία αποτελεσματική και ανταγωνιστική ε, άμυνα, όχι μόνο σε επίπεδο εμπορικό, αλλά και σε επίπεδο τεχνολογικό και σε επίπεδο ερευνητικό. Γιατί είναι γεγονός ότι ε, μπορεί να γίνονται περισσότερες έρευνες όσον αφορά το πολιτικό κομμάτι και θα ήθελα να επεκρετήσω την, να επενέσω τη δουλειά του κυρίου Έλερ στην Επιτροπή Ήτρε ως προς αυτό υπάρχει και το θέμα της στρατηγικής αυτονομίας και δεν είναι αυτό. Αν θέλουμε να θέσουμε έναν ακόμη αμυντικό λίθο ε, στο θεμέλιο της οικοδόμησης της αμυντικής βιομηχανίας, πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν είναι μόνο έμποροι κανονιών ε, η αμυντική βιομηχανία, είναι και ε, θέμα έρευνας, είναι και θέμα τεχνολογίας που ε, που είναι τομείς που έχουν εφαρμογές ε, και στο πολιτικό κομμάτι, όχι μόνο στο στρατιωτικό. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να το ξέρουμε αυτό και είναι κάτι το οποίο είναι μία αναστρέψιμο. Αν χάσουμε μία αμυντική τεχνολογία, δεν μπορούμε να την ξαναβρούμε και αυτό στοιχίζει και σε θέσεις εργασίας αλλά και σε οικονομική ευημερία. Το τρίτο μου ε, σημείο που έχει να κάνει με το θέμα αυτό της στρατηγικής αυτονομίας όλα τα κράτη-μέλη και μερικές φορές και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί που δεν ε, ε, σκέφτονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη στιγμή που πρέπει να εξοπλιστούν. Ίσως φαίνεται λιγάκι καρικατούρα όλο αυτό, αλλά η αμυντική ε, βιομηχανία είναι πολυεθνική για να το πω έτσι. Δεν είναι ότι είναι εθνικιστικό αυτό που λέω. Όταν ευρωπαϊκό όταν ευρωπαϊκό κράτο θέλει να εξοπλιστεί, καλύτερα είναι να βλέπει πρώτα τι υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και οι περισσότερε άλλε χώρε το κάνουν αυτό. Ακόμη και οι πιο φιλελεύθερε προστατεύουν κατά κάποιο τρόπο τι ε, ε δικέ του αγορέ και νομίζω ότι είμαστε λίγο αφιλεί ω προ αυτό το θέμα στην Ευρώπη. Και θα το δούμε στα επόμενα χρόνια ότι κάποιε χώρε ε, θα ακολουθήσουν προγράμματα εξοπλισμού αρκετά ε, ενδιαφέροντα και διαφοροποιημένα. Δεν σημαίνει υποχρεωτικά υποχρεωτικά ότι πρέπει να πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού να ψάξουμε τεχνολογίες που τις έχουμε στη διάθεσή μα εδώ στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Έλερ, ε, τέλος ε, ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο τη Επιτροπή Εξωτερικών Θεμάτων που είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε εδώ τη συζήτηση ε, σε ανώτερο επίπεδο, συζήτηση που γίνεται εδώ και καιρό στη ΣΕΝΤΕ και πολλοί ομιλητές ε, το θεωρούν χρήσιμο και σημαντικό. Δύο συγκεκριμένα παραδείγματα. Στην Ευρώπη δεν ε, παράγουμε ε, τεχνολογία στρατιωτική. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα τζιπ ευρωπαϊκό που να λειτουργεί με τη σημερινή τεχνολογία. Ευρωπαϊκή δεν υπάρχει τέτοια σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία. Όταν κάνουμε ένα joint call στο κέντρο διοίκησης και ε, παρακολούθησης, ε, μπορούμε να έχουμε συμπληρωματική δράση προς τα κράτη-μέλη και το ΝΑΤΟ. Δεν είναι επικάλυψη, δεν είναι διπλή δουλειά. Σε, ε, στο ίδιο επίπεδο θα πρέπει να κινούμαστε για τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου, command and control. να δούμε τι δυνατότητες έχουμε, τι ικανότητες έχουμε και βραχυπρόθεσμα τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό θα είναι το χρήσιμο. Τι ερευνητική δράση έχουμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλιώς κάνουμε μια οδυνηρή συζήτηση που μας πονάει και δεν προχωράμε γιατί αναλωνόμαστε σε αυτή την κρίνια. Ευχαριστώ πολύ. <coughs> Ευχαριστώ που κάναμε αυτή την πρώτη συζήτηση που δεν ήταν πρώτη συζήτηση. Κύριε Γκάλερ, κύριε Έλερ, σας ευχαριστώ που φέρετε τη συζήτηση εδώ. Μια σύντομη Ε, παρέμβαση για αυτά που είπε ο συνάδελφος Γκάλερ για τις επικαλύψεις και τις διπλές δουλειές. Τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένοι της Μεγάλης Βρετανίας, δίνουν 40 με 50% των ε, αμυντικών δαπανών στους Αμερικανούς. Γιατί δεν έχουμε αυτή τη συνέργεια, χάνουμε λεφτά, δεν έχουμε αρκετό προγραμματισμό, δεν έχουμε αρκετή κατανομή ε, επιμερισμό εργασίας και πάει λέγοντας και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Θα πρέπει να σταματήσουν οι Αμερικανοί να λένε ότι επικαλύπτουμε τον ΝΑΤΟ. Δυνατότητες δικές μας ε, θέλουμε να αναπτύξουμε, όχι να κάνουμε παράλληλη δουλειά με τον ΝΑΤΟ. Να σταματήσει αυτή η συζήτηση για το duplication. Είναι η συζήτηση του παρελθόντος αυτή. Ακόμα και οι Βρετανικές ενόπλες δυνάμεις και οι Γαλλικές ξέρουν ότι έχουν περιορισμούς και θα πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε κοινό σχεδιασμό, αμυντικές προμήθειες και έρευνα. Για να έχουμε ωφέλη όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. that point the chairman <laughs> Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του Προέδρου που άφησε την τελευταία του πνοή, λέει ο κύριος Έλε.